Präsident. Καλημέρα κυρίε και κύριοι. Άρχεται η συνεδρίαση. Περνάμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης, που είναι δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 20 και 21 Μαρτίου 2014. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Κούρκουλεκ, μέρος του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, το Ελληνό Συνέδριο παραδοσιακά αφιερώνεται ε, στην